Οι αρμόδιες λιθουανικές αρχές με ενημέρωσαν για την ε, εκλογή της κυρίας Λαΐμαν Ανδρικιένε από 30 Μαΐου 2016, η οποία και θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπέρκης. Καλώς ορίζω τη νέα συνάδελφο και να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεσμεύεστε και έχετε όλα τα δικαιώματα σε ό,τι